έξι ψηφίσματα για τις βίες διώξεις στο Ζιμπάμπουε. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, πόχες, κρίνονται. Επτά ψηφίσματα για την κατάσταση στην Καμπότζη. Ιδιαίτερα δε η περίπτωση δεν και πάλι υπάρχει κοινό ψήφισμα, το ψηφίζουμε υπέρ. Τα. χες. Γίνεται και αυτό. Και τέλος. Για τον Βόρειο Κάφικασο επίσης έξι ψηφίσματα. Την κατάσταση των δικαιωμάτων στο Βόρειο Κάφικασο και τις διώξεις κατά του Ολέγκορ Έχει ένα, υπάρχει ένα κοινό ψήφισμα, αλλά Υπάρχει μια προφορική τροποποίηση. Έτσι δεν είναι κύριε Μπόσελτ, μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφο Λατσπέργη που γνωρίζει σαν την τσέπη του το Βόρειο Κάφκασο ε, άφησε ε, μερικές μικρές προφορικές τροπολογίες που διευκρινίζουν το κείμενο και σα παρακαλεί να τον υποστηρίξετε. Θα τον εκπροσωπήσω εγώ και θα σα τι αναφέρω στο σημείο 3 αναγνωρίζει το δικαίωμα της Ρωσίας να καταπολεμήσει την πραγματική τρομοκρατία. Να μπει η λέξη πραγματική στην τρομοκρατία για να το διευκρινίσουμε. Διότι συχνά είναι πρόφαση η τρομοκρατία εκεί. Και στο πέμπτο θα θέλαμε να προσθέσουμε. Τονίζει ότι η συνεχιζόμενη ατιμορρησία, lasting να προσθέσουμε στο impunity. Και στο 15 θα θέλαμε να προσθέσουμε εκφράζει την απόρριψη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 η Νομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού,